Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς και συναδέλφισες, η χρονική ακρίβεια είναι προνόμιο των βασιλέων. Δεν είμαστε βασιλείς, είμαστε επιτροπή, αλλά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μια τροποποίηση στην μέση διάταξη, ό,τι αφορά τα θέματα της έγκρισης των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου προτείνεται να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία. Και αυτό έχει να κάνει με την διαθεσιμότητα των μελών, των υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να λάβουν υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και θα θέλαμε να ζητήσουμε και από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε στην νέα σε διάταξη. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Σόντεργα τώρα. Πρόκειται για την ειδική έκθεση 24-2012 για την ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του σεισμού στα Αμπρούτσι το 2009. Έχει ο εισηγητής ένα έγγραφο εργασίας και σήμερα λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Σέρον Σόντεργατ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος το πλαίσιο αυτής της συζήτησης νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ήταν ένα πολύ σοβαρό γεγονό. Ο σεισμό αυτό που έλαβε χώρα το 2009 οδήγησε στο θάνατο 300 ατόμων. Πολλά περισσότερα άτομα τραυματίστηκαν και ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι κατέστησαν άστεγοι ως εκ τούτου του σεισμού με στόχο να βοηθηθούν τα θύματα αυτής της τραγωδίας, το Νοέμβριο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει ένα σημαντικό ποσό 493, κάτι εκατομμύρια από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ήταν το πιο σημαντικό ποσό το οποίο δόθηκε ποτέ από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Και αυτό καταδεικνύει σε ποιο σημείο ήταν δύσκολη και σοβαρή κατάσταση μετά το σεισμό. Το θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτή τη συζήτηση είναι διτό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο τα ποσά αυτά τα οποία χορηγήθηκαν δαπανήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες. Και δεύτερον, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο τα θύματα της καταστροφής του σεισμού αυτού της Άκυλα είχαν επαρκή υποστήριξη από τα χρήματα αυτά που δόθηκαν. Αν υπήρξε αυτό το οποίο ονομάζουμε value for money στα ελληνικά, δηλαδή εάν έπιασαν τόπο τα λεφτά αυτά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέματα αυτού του είδους. Το είχαμε πράξει ήδη και μετά την ε, επίσκεψη της Επιτροπής μας στην Λάκουλα το 2010, όταν θέσαμε στην Κομισιόν μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία μας δημιουργούσαν ανησυχίες. Γιατί ήδη τότε είχαμε την εντύπωση ότι κάποια πράγματα δεν είχαν πάει καλά. Η έκθεσή μας μετά από αυτή την επίσκεψη του 2010 ζητούσε από την Κομισιόν και παραθέτω εδώ να προχωρήσει σε ένα λογιστικό έλεγχο ad hoc για το Ταμείο Αλληλεγγύης σε σχέση με το κόστος ανακουφιστικής βοήθειας και αποκατάστασης και σε σχέση με την κανονικότητα των συμβολέων, των συμβάσεων που συνήθισαν με τους προμηθευτές. Αυτό λοιπόν, κλείνω την παράθεση, αυτό είχε εκφραστεί ήδη μετά από την επίσκεψή μας το 2010 στην Λάκυλα. Το κατά πόσον είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για την ε, χορήγηση της βοήθειας αυτής. Διότι αυτή η βοήθεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για παραθέτω ανακοφιστική έκτακτη βοήθεια καθώς και στέγαση των σεισμοπαθών ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες του πληθυσμού που είχε πληγεί. Προσωρινή στέγαση και άμεσες ανάγκες των σεισμοπαθών. Το άρθρο 3 παράγραφος 2β του Ταμείου Αλληλεγγύης και πάλι σας παραθέτω αυτά που λέει πρέπει να δοθεί μια προσωρινή στέγαση και να χρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών. Τώρα, ένα άλλο σημείο το οποίο μας απασχολεί, κατά πόσο υπήρξε πλήρης και επαρκής έλεγχος για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να αποφευθεί μια αύξηση των τιμών και να αποφευθεί ότι ένα τμήμα των κονδυλίων τα οποία χορηγήθηκαν να πάνε στις λάθος τσέπες. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα και μάλιστα μπορούμε να το συζητήσουμε επί τη βάση της ειδική έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Και η Κομισιόν έχει συντάξει μια έκθεση η οποία είναι απόρριτη. Δεν μπόρεσα να, την, ε, να κρατήσω σημειώσεις για αυτά τα οποία περιείχε η έκθεση. Δεν μπορώ να παραθέσω στοιχεία αυτής της έκθεσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει λοιπόν βάση συζήτησής μας. Έχουμε όμως την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση μπορεί να είναι μια βάση για τα θέματα αυτά γιατί θέτει τον το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων μερικών πολύ σημαντικών στοιχείων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνει ακόμα και διαλαμβάνει όλα τα σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία προκύπτουν από αυτή την έκθεση. Κατάρχην, ένα μεγάλο μέλος της ε, αρρωγής χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν λιγότερο ε, μόνιμες λιγότερες ε, μόνιμες κατοικίες και περισσότερες προσωρινές <clears throat> κατοικίες. Και βάσει της έκθεσης οι τιμές των ακινήτων αυτών ήταν πολύ ανώτερες από τις τιμές 158 πάνω από την τιμή αγοράς, λέει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Και εδώ συνοψίζεται με λίγες γραμμές η άποψη του ελεκτικού συνεδρίου και θα τις παραθέσω γιατί στην Ιταλική ειδησεογραφία υπήρξαν κάποιες ε, παρεξήγησεις οι οποίες ανεφάνισαν. Είπαν ορισμένοι ότι το 158% είναι τα δικά μου στοιχεία, ότι εγώ δήλωσα ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά αυτά τα κονδύλια. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Εγώ απλώς μετέφερα αυτά τα οποία λέει το ελεκτικό συνέδριο. Αν θέλετε να επιτεθείτε εναντίον κάποιου, θα πρέπει να επιτεθείτε κατά του ελεκτικού συνεδρίου. Απλώς μετέφερα αυτά που είπε το ελεκτικό συνέδριο, που είπε ότι περίπου 30% 144 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν για δράσεις οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμες επί τη βάση του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο ΚΑΖΑ δεν ανταποκρίνεται στις ειδικέ προϋποθέσεις του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν ήταν χρήσιμο για να αντιμετωπίσει τις επιτόπιες ανάγκες. Δημιουργήθηκαν λοιπόν μόνιμες κατοικίες αντί να υπάρξουν προσωρινές κατοικίες. Το σχέδιο Καζά ε, καταδαπάνησε 350 εκατομμύρια ευρώ, 70% λοιπόν της συνολικής χρηματοδότησης και η στρατηγική η οποία χρησιμοποιήθηκε για το πρόγραμμα Κάζα κάλυψε τις ανάγκες 15.000 ατόμων οι οποίοι επλήρησαν από τον σεισμό αλλά δεν αντιμετώπισε τις συνολικές ανάγκες του πληθυσμού. Ήταν πιο πολύ δάπανες οι στεγάσεις βάσει του προγράμματος Κάζα από ότι η κανονική στέγαση, ενώ μια κανονική αξία ακίνητου οικίας. Και δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού πλήρως. Αυτά λέει το ελεκτικό συνέδριο σχετικά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να είμαι πιο επακρίβης για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να προτείνω η Επιτροπή μας να υποστηρίξει τα συμπεράσματα αυτά του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν είναι προσωπικά μου συμπεράσματα όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι συμπεράσματα στα οποία κατέληξα εγώ προσωπικά, είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το ελεκτικό συνέδριο. Και αυτό μας φαίνεται τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Δηλαδή, κατά πόσο τα θύματα του σεισμού έχουν τύχει επαρκή επαρκούς χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης και αν τα λεφτά αυτά έπιασαν τόπο. Και η απάντηση εδώ είναι σαφής, όχι. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. για, με το ποσό το οποίο δόθηκε ως αρρωγή. Δόθηκε, δημιουργήθηκαν καταλήματα για ένα τμήμα μονάχα, για ένα πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού που χρειαζόταν στέγαση. Ήταν ιδιαίτερα πολυδάπανα αυτά τα καταλήματα και ένα μεγάλο μέρος τους αντιμετώπισε και προβλήματα κατασκευαστικά και είτε υπήρξε αμέλεια και ανικανότητα στην κατασκευή υπήρξε και δόλος. Εγώ πήγα πολλές φορές στην ε, Λάκυλα μετά από το σεισμό. Ήμουνα και όλα στην ε, προηγούμενη Κυριακή και Δευτέρα. Πήγα στο σημείο αυτό, στο χώρο που αναφέρεται στην έκθεση, όπου δεν ξέρω πολύ καλά αν αυτός ο οικισμός κατασκευάστηκε στο Κάνσα αν ε, έχει χτιστεί με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο οικισμός είχε σαν στόχο να καλύψει τις ανάγκες μερικών εκατοντάδων σεισμοπαθών, αλλά κανείς δεν εκεί. Έχει εγκαταληφθεί αυτός ο οικισμός, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν ανθιυγιεινές αυτές οι εγκαταστάσεις στον οικισμό συνελήφθη ο υπεύθυνο για την κατασκευή αυτού του οικισμού και θα πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Αυτή δεν είναι μια μοναδική ιστορία εξάλλου. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις τέτοιες που αναφέρονται στην έκθεση και εγώ εντυπωσιάζομαι για το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν μπόρεσε να διακριβώσει επακριβώς τι ακριβώς συνέβη Ανεξάρτητα από όλα αυτά, το συμπέρασμά μας είναι το ίδιο. Έχει παραπλανηθεί ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, ο οποίος έδωσε χρήματα για να γίνει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ακόμα χειρότερα οι άστεγοι του σεισμού της ε, Λάκυλα και αυτοί ήταν θύματα παραπλάνησης γιατί δεν έλαβαν ποτέ τα χρήματα τα οποία έδωσε για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν πρέπει να έχουμε <clears throat> μια ιδιαίτερα επικριτική στάση. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα θέλαν να προχωρήσω ακόμα περισσότερο στις κριτικές μου έναντι της Κομισιόν και να ζητήσω την πλήρη ε, επιστροφή των χρημάτων αυτών από την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά εγώ προσπαθώ στα έγγραφό μου να έχω την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση σε σχέση με τα σημεία κριτικής. Παραμένω όμως τελείως ε, ανοιχτός, αν κάποιος μπορεί να μου υποδείξει κάποια διόρθωση σε αυτά τα οποία έχω γράψει με ανοιχτό σε οποιαδήποτε διόρθωση. Ε, νομίζω ότι το βασικό συμπερασμά μου που έλκεται από την εκθέση του ελεκτικού συνεδρίου είναι απόλυτα σαφέ. Θέλω και πάλι κλείνοντα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την ειδική του έκθεση που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και περιμένω την συνείδηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε, ε, συνάδελφε Σεντεργκάρτ, για την παρουσίαση του εγγράφου εργασία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ήτελε, μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου, που μας υπέβαλε την ειδική αυτή έκθεση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να καλωσορίσω τον ε, τον υποδιευθυντή του κ. Πόμπαντς ε, της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ανοίξει ο γύρος της συζήτησης Ποιος θέλει από πλευρά των βουλευτών να πάρει το λόγο. Δύο, τρει ζητούν το λόγο. Ο κύριος Ριβελίνη. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πω είμαστε ενώπιον μια κατά μέτωπο επίθεσης ε, κατά της Ιταλίας. Ο συνάδελφος μάλιστα έκανε μια συνέντευξη τύπου πριν να παρουσιάσει την έκθεσή του εδώ. Και πιστεύω πως χρειάζεται να αναλυθεί η τεκμηρίωση που λάβαμε τόσο από το ναι, ελεκτικό συνέδριο όσο και από την Κομισιόν ε, που η Κομισιόν σε σχέση με το ε, συνέδευξη τύπου του κ. Σόντεγκαρντ απάντησε με συγκεκριμένο τρόπο λέγοντας ότι το έγγραφο Σόντεγκαρντ φαίνεται να μην έχει συγκεκριμένη δομή και να είναι πολύ ε, περίπλοκο και υπάρχουν διάφορες παραλήψεις όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Άκουλα και τις πτυχές που σχετίζονται με τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Εμείς απορρίπτουμε κάθε, κάθε αναφορά σε ε, στην μη ε, σωστή παρακολούθηση, στη λάθος παρακολούθηση από πλευρά της Κομισιόν της κατάστασης. Ή σε σχέση με τα όσα μπορούμε να ξέρουμε εμείς, όλα τα ιταλικά θεσμικά όργανα ε, δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε συμμετείχαν σε κάποια, στη δημόσια κρόση που έγινε στις 26 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, όπου ήταν παρόντες ο δόκτωρ Ήταλ που, ήταν, που είναι παρόν και εδώ, ο κύριος Πόπενς ε, της DG Regio, ο πρόεδρος ε, της ε, περιφέρειας του Μπρούτζου, ο δήμαρχος της Άκουιλα, ο πρόεδρος της επαρχίας, ο Γενικός Διευθυντής της Πολεοδομίας, ο Γενικός Διευθυντής της Πυροσβεστικής, ο αρχηγός της πυροσβεστικής και εκεί θα μπορούσε να εκφράσει τις απορίες του και να αποσαφηνεί τις ιδέες του. Δεν το κάνει αυτό όμως με βάση στοιχεία τα οποία εμείς τώρα θα δούμε και θα αναλύσουμε. Ε, προέβησε σε συνέντευξη τύπου που μέχρι ότου μέχρι τι αποδείξεις του εναντίου και μέχρι, ε, και μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία απλά αμαυρώνει τη φήμη της Ιταλίας. Ορισμένα σημαντικά τώρα στοιχεία της έκθεσής του. Εκείνος ε, λέει πως υπήρξαν, ε, ε, υπήρξε δίδυση της μαφίας στην νοικοδόμηση και το λέει αυτό διότι πήρε μια φράση της κυρίας Όλγα Καπάσο από την Εθνική Διεύθυνση πολέμηση της Μαφίας. Ο κύριος Όντεγκαρ ξεχνά, ο, ίσως ξεχνά, ξεχνάει θέλημένα, ότι μια τέτοια δήλωση, αυτή η δήλωση μάλλον έγινε τους μήνες αμέσως μετά το σεισμό και αμέσως μετά την αρχή της ανοικοδόμησης και ο στόχος ήταν να μην διεισδύσει η μαφία στις δημόσιες συμβάσεις. Εγώ ε, ήμουν εισηγητής και στις 16 Μαΐου του ίδιου έτους ε, καταρχήν επισκέφθηκα την εισαγγελία της, ε, της Άκουιλα και την παρουσία μαρτύρων έλαβα την εξή απάντηση από τον εισαγγελέα σε συγκεκριμένο μου ερώτημα, ότι δεν υπάρχουν πέρα από μεμονωμένες ε, περιπτώσεις, δεν υπάρχει ε, σύστημα τύπου μαφίας ε, στην περιοχή. Το λέει και ο, ο ε, Περιφερειάρχης τον οποίο επισκεφθήκα επίσης ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται κατά της μαφίας. Το λέει επίσης ο κύριος Πόπερς κατά τη διάρκεια της ακρόασης που έγινε στις 26 Ιουνίου όπου ε, είπε ότι δήλωσε ότι δεν έχουν ε, ε, εντοπιστεί απάτες που μάλιστα είναι αρμοδιότητα της Όλαφ και που δεν ξεκίνησε καμία σχετική διαδικασία δεν, υπήρξε, δεν εντοπιστεί και λοιπόν καμία περίπτωση όπου να μπορούσε κανείς να υποψιαστεί την ύπαρξη διείσδυση της μαφίας. Ο κύριος Όντεργα μιλά για υποθέσεις για, για ε, σπίτια τα οποία δεν είναι προσωρινά αλλά μόνιμα και έτσι ε, αλλοιώνει τα λόγια του Δημάρχου της Άκουιλα που στις 26 Ιουνίου είπε ότι η ε, ανοικοδόμηση θα διαρκέσει 8 με 12 χρόνια και αντίθετα στην έκθεση Σόντεργαρντ η φράση 8 με 12 χρόνια του, του Δημάρχου ε, έχει αλλάξει και αναφέρεται ως 25 ετία. Διπλασιάζει δηλαδή το χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο ποτέ δεν είπε ο, ο Δήμαρχος. Επιπλέον λέει ότι όλα τα σπίτια που κατασκευάστηκαν, κατασκευάστηκαν με πολύ κακή ποιότητα. Και χωρίς όμως να γίνει καμιά γνωμάτευση, καμιά ειδική μελέτη. Και φέρνει κάποιες ε, παραδείγματα τα οποία υπήρξαν. Είναι 94 άνθρωποι στο χωριό Κανταμέσα, 45 σε ένα άλλο χωριουδάκι και 15 σε ένα παραάλλο. άλλο. 154 άνθρωποι από ένα σύνολο 48.800 εκτοπισμένων. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι όλα τα αντισυσμικά συστήματα είναι εκτός, είναι παράνομα. Η Κομισιόν λέει πως μόνο το 2,5% από τα αντισυσμικά συστήματα δεν είναι απόλυτα κατάλληλα. Όχι ότι έγιναν παράνομα ή εκτός των ε, προδιαγραφών, ε, αλλά απλώς ε, δεν, έχουν, δεν είναι απόλυτα σύμμορφα με τις δια, αντισυσμικές διατάξεις. Άρα ο κ. με βάλει και εδώ. Εδώ μάλλον δεν θα είδατε και τα... Τα 12 εκατομμύρια προγράμματα έγιναν από πλευράς των Ιταλικών αρχών. Επιβεβαιώνει επίσης πως η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανώτερη, είναι, ε, υπερβολική, ε, εκτός δηλαδή των ε, κανονικών και συνηθισμένων ορίων. Ο κύριος Σόντριγκαρντ όμως ίσως να μπορούσε να διαβάσει την σχετική έκθεση και να δει πως εκεί έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες για 919 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Δηλαδή, 350 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντός των κοινοτικών κανόνων. Λέει πως ε, τα σπίτια κόστησαν 158% παραπάνω, αλλά δεν θυμάται τις κλιματικές, γεωγραφικές συνθήκες ε, δεν γνωρίζει ίσως την Άκουιλα που είναι μία από τις 20 ευρωπαϊκές χώρες τέχνης. Πρέπει να αποκατασταθεί όπως ήταν. Δεν μπορεί δηλαδή να τα γκρεμίσει όλα και να τα φτιάξει όπως να είναι. Και είναι σαφέ πως αυτή η κατάσταση οδήγησε σε ένα ψηλότερο ποσό, αλλά αυτό πιστοποιείται και έχει δοθεί το πράσινο φω από την Κομισιόν. Κάνει λόγο επίση ε, για το ότι έγιναν δαπάνε υπερβολικέ για τους ε, πυλώνες ε, τους ατσάλινους και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τσιμεντένιοι πυλώνες. Δεν ε, λέει όμως ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι ατσάλινοι οι τσιμεντένοι πυλώνες εκεί που χρειαζόταν και εκεί όπου λόγω χρονικών περιορισμών ή για τεχνικούς περιορισμούς χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν άλλου είδου πυλώνες, δηλαδή ατσάλινοι, εκεί και όντως χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό που με λυπεί λοιπόν με τον συνάδελφο Ζόντεργαν είναι ότι μέχρι σήμερα δεν μας έδωσε εμπειρογνωμοσύνε, δεν μα έδωσε γνωματεύσεις, δεν μα έδωσε χαρτιά. Εμείς διαβάζουμε μόνο ούτε πλάνα, ούτε σχέδια, ούτε χάρτες. Μας έδωσε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και της Κομισιόν που λένε άλλα από αυτά που λέει ο Ζόντεργκαρντ. Αν διαβάσει κανείς αυτά τα χαρτιά, το 2,5% δεν σημαίνει το σύνολο. Δεν μπορεί λοιπόν να μας λέει ότι όλα έγιναν με αρνητικό τρόπο. Αυτή η Διαφήμιση βεβαίως το ξέρω γιατί όταν εγώ ορίστηκα εισηγητή για το ΕΛΚΑ και καταρχήν πήγα στι 16 Μαου και επισκέφθηκα όλα τα θεσμικά όργανα, την εισαγγελία, την, ε, το ελεκτικό συνέδριο, το τμήμα της Πολεοδομίας, το δήμαρχο της Άγουλα, τον πρόεδρο της ε, επαρχίας και της περιφέρειας και τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όταν λοιπόν ε, εκεί επί επιτόπου ε, όλοι αυτοί συναντιόνταν θα είχα πραγματικά φωνάξει ε, αν μιλούσε για σκάνδαλο και θα είχα ακροαματικότητα τεράστια. Σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου θα με είχαν βγάλει. Αλλά δεν το έκανα προς το συμφέρον της κοινότητας και θα διαβάζουμε ένα σωρό πράγματα και πριν να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις, ας δείξτε μας χαρτιά, δείξτε μας Στι εμπειρογνωμοσύνης δεν μπορείτε να μου λέτε πως 154 πολίτες που χρειάστηκε να αλλάξουν σπίτι γιατί το σπίτι τους ε, ε, είχε κρυφθεί ακατάλληλο μπορούν να συγκριθούν με τους 48.800 εκτοπισμένους πολίτες λόγω εκείνου του σεισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ελπίζω πως με τον συνάδελφο Σόντεργα θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε γιατί αν έχει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχω εγώ θα κάνουμε μαζί όλους τους αγώνες και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ε, ε, φανεί η αλήθεια. Αν όμως δεν έχει άλλη εμπειρογνωμοσύνη να μας δώσει, τότε θα πρέπει να τη διαβάσει σωστά, χωρίς να την παραποιήσει και να μην ε, ε, λασπολογή για μια δουλειά τέτοια αποκατάσταση που δεν εξυπηρετεί ούτε τους ε, κατοίκους της Άκουλα, ούτε τους Ιταλούς, ούτε και τους Ευρωπαίους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ράγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκάιρ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σόντρεγκάρτη για το έγγραφο αυτοεργασίας. Ε, που έχει, για το θέμα αυτό που έχει απασχολήσει πολύ την Επιτροπή μας. Ένα ταξίδι, μια αποστολή επιτόπου έχει δραγματεί και όντως ανησυχούμε κάπως ότι η συζήτηση γίνεται πολύ συναισθηματική, υπερβολικά ίσως και απομακρύνεται από το πυρήνα του θέματος το οποίο καλούμαστε να εξετάσουμε. Το θέμα λοιπόν ε, της προσβολής της Ιταλίας δεν είναι αυτό που μας απασχολεί και θα καλούσα να είμαστε λίγο λιγότερο συναισθηματικοί. Μιλάμε για ένα έγγραφο εργασίας. Το τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει συστάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ε, χορήγηση απαλλαγή ή όχι. Αυτό θα το ψηφίσουμε, αλλά το έγγραφο αυτό σκοπό έχει στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει ε, με τους ευρωπαϊκούς πόρους και όχι φυσικά να προσβάλλει μια χώρα. Και να σας υπενθυμίσω ότι αν ε, υπήρχε τέτοια υπόνοια θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την πολιτική του κατονομάζει του υπεύθυνου. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα που μας απασχολεί στην παρούσα φάση. Όταν λέει ο συνάδελφος ε, Ριβουλίνη ότι υπάρχει κάποια ραντασμένη ε, εκτίμηση κάποιων σημείων, στην, στο έγγραφο εργασία, θα ήθελα να επισημάνω ότι απλά υπογραμμίζονται σημεία τα οποία υπογράμμισε η Όλαφ και στα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Αυτό το γεγονός λοιπόν ότι δεν βρήκε ο κύριος Ριβελίνη να υπάρχει απάτη δεν είναι ότι όλα αυτά βρήκε στοιχεία. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε απάντηση από την ΟΛΑΦ. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό για την αξιολόγηση. Και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν κράτη όπου με τις πληροφορίες της κάθε υπηρεσίας ε, και με την αξιολόγηση αυτών είμαστε ή δεν είμαστε ικανοποιημένοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που λάβατε εκ μέρους της ε, ομάδας να μας δοθεί μία αναφορά από την περιοχή. Αλλά κανονικά δεν μας αρκεί αυτό ως απάντηση, το τι το λένε δηλαδή οι τοπικές αρχές. Ξέρω από τις μαφιόζικες πρακτικές ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν θύματα, ανθρώπινες ζωές. Μία κανονική πρακτική της μαφίας είναι ότι δίδεται ε, μία σύμβαση σε μία τέτοια εταιρεία η οποία πληρώνεται, αλλά τελικά παρέχει λιγότερε υπηρεσίε. Δεν ισχυρίζομαι ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά ούτε ο κ. Σόντερκατ λέει κάτι. Λέει ότι για τα χρήματα, τους πόρους που δαπανήθηκαν, τα κονδύλια που δαπανήθηκαν, είναι λιγότερες οι υπηρεσίες που τελικά χορηγήθηκαν. Δεν λέω ότι υπάρχει πραγματικά ε, συμπεριφορά μαφίας, ούτε όμως η έκθεση το λέει αυτό. Και ε, σε, αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε τι ευκαιρίες τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να πει ότι αυτό ισχυρίζονται οι τοπικές αρχές. Η δεύτερη μέθοδος, η δεύτερη δυνατότητα που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το φροντίσαμε και εμείς ως Επιτροπή είναι να ασχοληθεί η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το πράττει και θα αναμένουμε Αναμένουμε στην παρούσα φάση το αποτέλεσμα. ορίζω λοιπόν ε, το έγγραφο και θεωρώ ότι οι συστάσεις του εγγράφου σε καμία περίπτωση δεν ε, καταδικάζουν, δεν είμαστε σε δικαστήριο εδώ, δεν χρειαζόμαστε αποδεικτικά στοιχεία κατάρτισε ο συνάδελφο μια πολιτική έκθεση. Αυτό και έκανε και καλωσορίζω την έκθεση αυτή και θα δούμε τι θα γίνει στη συζήτηση για τη χορήγηση της απαλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιρενχάουζερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ είπε πάρα πολλά από τα οποία ήθελα και εγώ να αναφέρω. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα που δημιουργεί συγκινησιακές αντιδράσεις, πρόκειται για μια μεγάλη φυσική καταστροφή και δεν είναι παράξενο το ότι υπάρχουν συναισθηματικές αντιδράσεις. Παντός θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένο το έγγραφο του κ. Σόντεργατ και νομίζω ότι και τα σημεία επίκρισής του είναι τεκμηριωμένα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κύριε Ριβελίνη επιτίθεστε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Σόντεργατ. Εδώ δεν είναι ένα θέμα εθνικιστικών αντιπαραθέσεων, δεν είναι κάτι που αφορά ένα κράτος μέλος. Είναι απλώς μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συνέβη σε αυτήν την περίπτωση και να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό προσπάθησε να το κάνει ο κύριος ε, Σόντεργατ. Για μένα δεν υπήρξε αρκετή αναφορά στην έκθεση του ελεκτικού συνέδριου. Το ελεκτικό συνέδριο είναι αυτό το οποίο είπε ότι ήταν 158% ακριβότερα τα κτίρια τα οποία δημιουργήθηκαν και στα πλαίσια αυτού του σχεδίου Κάζα αναφέρθηκε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ότι κάποια από τα οικήματα τελικά δεν έχουν κατασκευαστεί. Όλα αυτά είναι περιεχόμενο της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Δεν νομίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να επιτεθεί κατά της Ιταλίας. Ίσως και το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να απαντήσει τώρα στο ερώτημα αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει για το ελεκτικό συνέδριο ένα προσωρινό οίκημα, ένα οίκημα ανάγκης, ένα κατάλημα ανάγκης. Πώς καθορίζει το ελεκτικό συνέδριο την έννοια αυτή της στέγασης έκτακτης ανάγκης Επίσης δεν έχουμε κανένα κανονισμό για το τι γίνεται με τα οικήματα τα οποία κατασκευάζονται. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια μνήα στα θέματα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα πάντα να ενοικιαστεί ένα οίκημα που έχει κατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί στην αγορά. Η κυρία Γκρέσλε και μετά θα ακούσουμε τα μέλη του Εκτικού Συνεδρίου και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα θέλετε να απαντήσετε. Η κυρία Γκρέσλε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ, να αναφέρω και εγώ κάποιες ερωτήσεις που έχω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έναν έλεγχο από τις 13 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2012 στην Ακουιλά. Και από την έκθεση αυτή προκύπτουν διάφορα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανάθεση των έργων. Και ξέρουμε πώς λειτουργούν τα αρθρωτικά ταμεία. Νομίζω ένα τρίτο όταν ε, μιλάμε για τέτοια ε, προβλήματα και ανάκτηση πόρων. Η επιστροφή πόρων στο 1 τρίτο. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, προσπαθήσατε να ελέγξετε τα ελαττώματα που υπήρχαν σε ό,τι αφορά τις οικοδομές ε, και πρόκειται να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα να αντιευκρινιστούν αυτέ οι κατηγορίε που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασία. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα, υπήρχαν τέτοιε ακατοματικέ οικοδομέ. Ενδιαφέρον ήταν αυτό που αναφέρει το έγγραφο εργασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση των υστέρων στο Άκουιλα για την όλη ιστορία. Υπήρχαν λοιπόν τέτοια ερωτώματα. Κατά δεύτερον, το έγγραφο εργασία προσδιορίζει ότι ένα τμήμα των εταιριών που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς και κέρδισαν τους διαγωνισμούς δεν έχουν πιστοποιητικό κατά της μαφίας. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πιστοποιητικό αυτό κατά της μαφίας παίζει ρόλο για την ε, ανάθεση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Το ελέγξατε αυτό. Ύστερα, σημαντικό θα ήταν να τοποθετηθεί η Όλαφ σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τα μέσα και να δούμε πότε θα κληροκριθούν όλα αυτά. Να μας μιλήσει όλα αυτή την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να διευκρινίσουμε, εγώ επισκέφτηκα και εγώ την Λάκουιλα, να διευκρινίσουμε η Ιταλία πόσα έδωσε μετά τον σεισμό. Θυμάμαι μετά από μια συζήτηση που δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί του ποσού που δαπάνησε η Ιταλία για την Λάκουιλα. Γιατί με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πολύ κατά πόσον τηρήθηκαν οι δεσμεύσει και περιλαμβάνονται στις συστάσεις. Έχω κάποια προβλήματα με κάποιες συστάσεις, γιατί δίδεται η εντύπωση ότι συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία